για την έκταση πρόοδου στην ανανεώσιμη ενέργεια και έκταση εφαρμογή σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση του κ. Μάρκου Πίπερ. Και το λόγο παίρνει η συνάδελφο Λόπε Περμέχιο ω εισηγήτρια για να ξεκινήσει. Για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αξιότιμοι σκιώδη εισηγητέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Δύο μήνες και κάτι πέρασαν από τότε που για πρώτη φορά καταθέσαμε το σχέδιο εκθέσεώς μας για την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες αλλά και τη Γραμματεία για την ταχύτητα και την προθυμία τους έτσι ώστε σήμερα να ψηφίσουμε. Χαίρομαι για την ε, μεγάλη σε πολλά σημεία παρόλο που δεν ήταν πλήρη συμφωνία τελικά στην τελική ψηφοφορία της Επιτροπής το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσανατολίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση των χωρών που δεν θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για το 2020 για το στόχο των ανανεώσιμων. Θα πρέπει όμως επίσης να προετοιμάσουμε την πρόταση για μια νέα οδηγία ανανεώσιμων μέχρι το 2030 που να διατηρεί τους δεσμευτικούς στόχους και να τους ενισχύει έτσι ώστε να πληρωθούν υποχρεώσεις καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής που συνήθισαν στην COP21. Τα ίδια λέει και η έκθεση Πίπερ για την ενεργειακή αποδοτικότητα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ συνάδει με τις οικονομίες, με την ενεργειακή απόδοση και προσκρούει στα ίδια εμπόδια στα κράτη-μέλη. Στόχος μας λοιπόν είναι να προωθήσουμε μία ενεργειακή μετάβαση προς ένα πιο οικολογικό, πιο δημοκρατικό και πιο κυρίαρχο μοντέλο απέναντι στα συμφέροντα των μοπολίων και των ολιγοπολίων που σήμερα κυριαρχούν. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε στον Επίτροπο κύριο Άρια Κανιέτε ποιες είναι οι πολιτικές που επηρέασαν πιο ανητικά τις ανανεώσιμες η κυβέρνησή του, στην οποία συμμετείχε και όλα τις έχει εκτελέσει. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα συστήματα πρόθεσης ΑΠΕ είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα και έρχονται απέναντι ε, στις ε, πιο βλαβερές μορφές ενέργειας. Η υποστήριξη των ΑΠΕ Χρειάζεται νέε επενδύσεις στη ε, διάδοση και στη μεταφορά μάλλον της ενέργειας. Υπάρχουν ε, προβλήματα για το περιβάλλον από άλλε μορφές ενέργεια. Υπάρχουν εναλλακτικέ που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι το φυσικό αέριο ή η πυρηνική ενέργεια. Οι ε, ΑΠΕ είναι αποτελεσματικότερες και πιο ανταγωνιστικέ. Θα πρέπει να έχουμε μηχανισμού παραγωγή ενέργεια που να ελέγχουν ε, τα μεγάλα ολιγοπόλια απέναντι. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε το δικαίωμα στην αυτοκατανάλωση και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς δημόσιου προγραμματισμού και ε, συμμετοχής στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και τα συλλογικά συστήματα παραγωγής, ε, διανομής και αποτελεσματικότητας στην ενέργεια. Και εδώ μιλώ και για την ηλεκτρική ενέργεια και για την ψήξη και για τη θέρμανση. Πιστεύουμε ότι στο παρελθόν η οδηγία υπήρξε χρήσιμο εργαλείο. Καλά, μπορεί να είχαν και κάποιε ανεπιθύμητε συνέπειες όλα αυτά που πρέπει να διορθωθούν, κυρίως σε ό,τι αφορά την παγκόσμια βιωσιμότητα και τη βιοενέργεια. Είτε είναι η βιομάζα ε, για ε, θέρμανση ή το βιοδίζελ για μετακίνηση, για καύσιμο. Το να είναι ανανεώσιμη η πηγή ενέργεια δεν σημαίνει ότι γίνεται σωστή χρήση. Ε, όπως βλέπουμε υπάρχει ανταγωνισμό στη γεωργία για παραγωγή τροφίμων ή καυσίμων και γενικότερα άλλα προβλήματα. Τελειώνω. Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μόνο τεχνολογική πρόκληση, αλλά και κοινωνική πρόκληση. Επειδή ε, λέμε και σε μια τροπολογία που πιστεύουμε ότι θα εγκριθεί, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια άναρχη μετάβαση που να μειώνει τις εργασιακές προδιαγραφές ή να υπονομεύει τη δημιουργία θέσεων ε, εργασίας στην ενέργεια. Γι' αυτό στην Ένωση τονίζουμε ότι θα πρέπει να προχωρούμε χέρι-χέρι με τους κοινωνικούς εταίρους για να ορίσουμε το νέο κοινωνικό, το νέο ενεργειακό μάλλον μοντέλο και να καταπολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Μόνο έτσι και με κοινωνικέ εγγύσει θα βοηθηθούν και τα φτωχά νοικοκυριά που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικό δικαίωμα που είναι αυτό στην ενέργεια. Ελπίζω στη συζήτηση να χτίσουμε γέφυρε και να βρούμε πλειοψηφία γιατί είναι πολύ μεγάλη σημασία του θέματο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ συνάδελφε Λόπε Περμέχη και τώρα έχουμε τον δεύτερο εισηγητή, ο κύριο Μάρκο Πίπερ για τέσσερα λεπτά. Επίση ευχαριστώ πολύ Πρόεδρα. Κύριε Επίτροπε, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, διεξάγεται το Βρετανικό Δημοψήφισμα και το θέμα λοιπόν εκεί, το θέμα είναι η αλληλεγγύη, η μείωση της γραφειοκρατίας και όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι μια κατάσταση διπλού ωφέλους, win-win και για το περιβάλλον. Η ενεργειακή αποδοτικότητα σημαίνει λιγότερη έκκληση βλάβερων ουσιών διοξιδίου του άνθρακα και πιο πολύ ενεργειακή αποδοτικότητα σημαίνει και λιγότερο κόστο. Για την ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή αποδοτικότητα σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια παροχή. Ε, γι' αυτό λοιπόν η οδηγία πρόκειται. Για την οδηγία αυτή επενδύουμε στο μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ε, το αντιμετωπίσουμε σωστά, τα αποτέλεσματα είναι σωστά. Μέχρι το 20%, μέχρι το 2020 θα πετύχουμε 20% μείωση τη ενεργειακή κατανάλωση, αλλά δεν ε, τίθεται θέμα σωστής εφαρμογής ε, της οδηγία, αλλά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιορισμένη κατανάλωση της ενέργειας. Ε, ο ενεργειακό ε, ισολογισμός της Ένωσης είναι μεγάλο επιτεύγμα, γιατί είμαστε παγκόσμιος πρωταθλητής ό,τι αφορά στις ΑΠΕ και σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά οι πολίτες, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα. Καταρχάς, ε, οι τιμέ, είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο. Και εδώ φαίνεται ότι αποδίδουν σιγά σιγά οι αποζημιώσεις για την παραγωγή ενέργειας και τη χορήγηση στην, ε, στο δίκτυο. Οι επενδύσεις, ε, ωστόσο, αποδίδουν κατά τρίτον. Έχουμε τη γραφειοκρατία, οικοσχεδιασμός, επισήμανση, ETS, μείωση των ε, καυσαερίων, η οδηγία για τα κτίρια. Φυσικά κάθε νομοθεσία έχει το λόγο ύπαρξή τη, ναι. αλλά να μην ξεχνάμε και αμελούμε ποιε είναι οι παράπλευρε συνέπειε ό,τι αφορά και τι ενεργειακέ πολιτικέ των ε, εθνικών κρατών μελών. Γιατί ε, προκύπτει μεγάλη γραφειοκρατία, αλλά τίθεται και το θέμα της, των πιστοποιητικών εκπομπών, γιατί ουσιαστικά τιμωρούμε για τα λάθη μας και τις επιχειρήσεις με πολύ μεγάλο νέο κόστος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό κυρίε και κύριοι. Για παράδειγμα το έθιξα αυτό στην ε, οδηγία για την ενεργειακή επενδυτικότητα και χαίρομαι πολλά, ότι πολλά από τα στοιχεία αυτά παρέμειναν σε ό,τι αφορά μεγαλύτερη καινοτομία για την αποδοτικότητα και όχι να κοιτάμε πάντα την εξοικονόμηση να παραμείνει ευέλικτη η οδηγία, προκειμένου να έχουν περιθώριο προσαρμογή στα κράτη-μέλη και σε ό,τι αφορά η, την ανάγκη ε, ομοιογενούς εφαρμογής των στοιχείων αυτών. Τονίσετε στην έκθεση. Συμφωνούμε σε αυτό στο Κοινοβούλιο, αλλά αυτό που δεν με βρίσκει σύμφωνο είναι μια οδηγία για εξοικονόμηση 40%. Υποχρέωση για την κατανάλωση ενέργειας. Εδώ το θέμα δεν είναι η αποδοτικότητα, το θέμα είναι η απαγόρευση ουσιαστικά χρήση ενέργεια, κυρίε και κύριοι. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε αν τα πήγαινε πολύ άσχημα η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κατανάλωση. Αλλά τα δεδομένα και τα στοιχεία είναι πολύ διαφορετικά. Έχουμε μειώσει πολύ την κατανάλωση και έχει αυξηθεί το ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια και έτσι λοιπόν έχουμε 25% λιγότερες ε, έκκληση βλαβερών ουσιών και έχουμε 50% μεγαλύτερη απόδοση. Είμαστε πάρα πολύ αποδοτικοί. Όποιο λοιπόν υποστηρίζει αυτό το 40% περιορισμό της χρήσης ενέργειας, νομίζω ότι αγνοεί αυτά τα πραγματικά γεγονότα. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ κατεπηγόντως τους συναδέλφους από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και από τους Φιλελεύθερους να ε, υποστηρίξουν τις τροπολογίες μας για την ε, γενικότερη κατεύθυνση μείωσης 30 κατά 40%, όχι όμως για την υποχρέωση ε, μείωσης κατά 40%, γιατί καταρχάς θα θέλαμε να δώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι πρώτα σε ό,τι αφορά την ε, μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συναδέλφους μου. Σας ευχαριστώ και τώρα τον λόγο έχει ο Αρίας Κανέτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, νιώθω μεγάλη μου χαρά που σήμερα βρίσκομαι εδώ και έτσι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τι γίνεται για ένα από του πιο βασικού πυλώνε τη ενεργική μα ε, πολιτική και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Και επίση θα πρέπει κάτι άλλο να, να δούμε το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο που παίζουν αυτοί οι άξονε τη πολιτική μα για του στόχου που έχουμε θέσει και τους στόχους της συνάντησης κορυφής του Παρισιού. Θέλουμε τώρα να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση της σχετικής πολιτικής. Ε, και αυτό θα γίνει το δεύτερο ημίση του έτους. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τους δύο συγητές γιατί ήταν εξαιρετική εργασία που έκανε για αυτές τις δύο εκθέσεις. Πρώτα πρώτα ε, για την έκθεση Πίπερ. Όπως γνωρίζετε, τώρα ετοιμάζουμε την αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών για ε, την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια. Και αυτό που θέλουμε τώρα είναι να θέσουμε κάποιους ε, στόχους και να τους πετύχουμε το 2030. Και γι' αυτό έχουμε ένα πλαίσιο και τα, πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα μέτρα. Και επίσης να εστιάσουμε προσοχή μα στο τι γίνεται στα κτίρια και να δώσουμε προτεραιότητα στους ε, κλάδους που μπορούμε καλύτερα να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Έχουμε κάποιες, ε, κάποια συμπεράσματα θα τα λάβουμε υπόψη για την αναθεώρηση που σας προανέφερα και συμφωνώ 100% με το συμπέρασμα έκθεσης Πίπερ ε, ότι θα πρέπει δηλαδή συστηματικά να ακολουθούμε την αρχή ότι πρώτα πρώτα θα πρέπει να υπάρχει ε, ενεργειακή απόδοση γιατί χρειαζόμαστε έναν στόχο ξεκάθαρο το 2030, κάτι το οποίο να το αγκαλιάσει η νομοθεσία, άρα προς τους επενδυτές και τους νομοθέτες να είναι σαφές το μήνυμα και έτσι να έχουμε τέτοιες μακρόπνοες επενδύσεις που να βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους. Αλλά αυτή η αναθεώρηση της πολιτικής μας χρειάζεται και άλλα πράγματα πέραν αυτού του στόχου. Θα πρέπει στα σοβαρά να εφαρμόσουμε την κείμενη νομοθεσία. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί η οδηγία της ενεργικής απόδοσης και το άρθρο 7, εκεί που λέμε για την υποχρέωση της εξοικονομίας ενέργειας και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αγκαλιάσουν αυτή την πολιτική με σοβαρότητα και να υπάρχουν κάποια συστήματα ελέγχου, επαλήθευσης και να γίνονται οι εξοικονομήσεις που χρειάζεται με στόχο το 2020. Οπότε το σχετικό άρθρο μπορεί να μας οδηγήσει στο 50% της που προβλέπει η οδηγία. Να έχουμε έτσι ένα εργαλείο αποτελεσματικό και να ευθυγραμμιστούμε ε, με το πλαίσιο που έχουμε τάξει για το 2030 και έτσι να μπορέσουμε ε, να έχουμε τη μείωση των ε, εκπομπών όπως απεφάσισε το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε τις δυνατότητες με τα κτίρια να έχουμε ενεργειακή απόδοση και ε, εξοικονόμηση να ε, είναι πιο φθηνή η ενέργεια και να προστατευτεί και η υγεία. Οπότε ιδίω όσον αφορά την νομοθεσία και τα κτίρια θα τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ τον εισηγητή που έλαβε υπόψη αυτά τα ζητήματα στο κείμενό του οπότε και θα συνεργαστούμε για αυτές τις νομοθετικές προτάσεις όλα αυτά βεβαίως ισχύουν και για την ε, οδηγία για τα ανανεώσιμα. Είναι μια οδηγία που έχει λειτουργήσει εύρυθμα και έχουμε αυτό το 16% εξοικονόμηση ε, το 2014 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλειοψηφία των κρατών μελών προχωρούν ολοταχώς προς την επιτύχηση των του 2020 και όλες οι χώρες πλην μιας ε, έχουν υπερκαλύψει το πλάνο και τους στόχους για το 2020 οπότε και εμείς μπορέσαμε να μειώσουμε τις ε, εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και να προχωρήσουμε όσον αφορά τα ανανεώσιμα. Παρ' όλα αυτά, κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να είναι στο ύψος ε, αυτής της έντονης προσπάθειας για τα επόμενα χρόνια, οπότε και εμείς έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας στην εφαρμογή της οδηγίας για τα ανανεώσιμα, κάτι το οποίο και για το Κοινοβούλιο ξέρω ότι είναι σημαντικό. Ε, Βεβαίω και όπω λέει και η έκθεση, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται μετά το 2020. Οπότε η αναθεώρηση τη οδηγία για τα ανανεώσιμα θα είναι ο πυλώνα, ο κεντρικό άξονα για αυτέ τι προσπάθειε. Να δούμε τι θα γίνει και με την αγορά τη ηλεκτρική ενέργεια και την πρωτοβουλία για την ε, διακυβέρνηση. Και θέλουμε να έχουμε ένα στεγανό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να πείθει του ε, επενδυτέ όσον αφορά την μεταρρύθμιση τη πολιτική μα και για τα ανανεώσιμα, για την ηλεκτρική ε, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, όλα αυτά θα είναι βασική λόγοι ούτως ώστε να ελκύσουμε επενδύσεις για τα ανανεώσιμα και έτσι η Ευρώπη να είναι ο πρωταθλητής σε αυτό τον ε, τομέα. Με την ανθεώρηση της οδηγίας λοιπόν θέλουμε να καλύψουμε τις ανησυχίες που εσείς εκφράζετε ή στις τροπολογίες τι θα γίνει δηλαδή όσον αφορά την ψήξη και την θέρμανση και για το τι θα γίνει με τον καταναλωτή. Ε, θα πρέπει να υπάρξει λιγότερη γραφειοκρατία και πιο ελαφρύ θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Οπότε ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία αλλά και τους στόχους που έχουμε τάξει το 2020. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν και οι εθνικοί στόχοι το 2020 και αυτοί οι στόχοι να είναι η αφεντηρία. Έχουμε επίσης τρεις τομείς ε, που θα μας βοηθήσουν για ε, αυτούς τους στόχους μεταφορές, ε, ψήξη, θέρμανση, εξηλεκτρισμός ε, για κυρίως να προσέξουμε τις μεταφορές επίσης σημαντικό είναι το τι θα γίνει με τις ανώσιμες πηγές ενέργειας και οπότε θα πρέπει η αλλαγή αυτή να παγιωθεί και να υποστηρίξουμε τις εθνικές προσπάθειες και όπως προανέφερα προχωρούμε προς καλύτερο σχεδιασμό της αγοράς ε, εμπορία των εκπομπών και έτσι αυτοί που παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια να διευκολυνθούν. Τέλος, στην έκθεση είδαμε ότι έχουμε κάποια κριτήρια βιωσιμότητας για την βιοενέργεια, τα οποία δημιουργούν μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλουμε τέτοιου είδους πολιτική βιωσιμότητας για βιοκαύσιμα και βιομάζα που παράγουν ε, ε, ανανεώσιμη ενέργεια και θεωρούμε ότι έτσι ε, είμαστε ρεαλιστές, αντιμετωπίζουμε τις ε, εκπομπές, προστατεύουμε το περιβάλλον και προσπαθούμε να εξαλείψουμε την ε, γραφειοκρατία. Κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσω τονίζοντας το ότι είναι αυτή η συζήτηση πολύ σημαντική, όπως και η συμβολή του Κοινοβουλίου για να προετοιμάσουμε τις μέλουσες νομοθετικές προτάσεις και έτσι θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε, να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε τάξει. Θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τους επενδυτές και το ΕΦΣΙ για τις στρατηγικές επενδύσεις μας έδωσε κάποιες δυνατότητες. Θα πρέπει να φανούμε έξυπνοι και να το εκμεταλλευτούμε για να εμπλακούν περιφερειακές αρχές, τοπικές αρχές για να αξιοποιηθεί αυτό το εργαλείο. Ε, Κατακλείδη σας αναφέρω ότι ευχαριστούμε ε, θερμά για αυτές τις δύο εκθέσεις και σας ε, διαβεβαιώνω ότι στις επόμενες ε, νομοθετικές μας προτάσεις θα είμαστε φιλόδοξοι και η αποτελεσματικότητα της ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση θα ακολουθεί τόσο που αποφασίσαμε στο Παρίσι για τον άνθρακα και τους άλλους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε Άρια Και τώρα ακολουθούν οι συνάδελφοι εξ ονόματος των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Πρώτη κυρία Πετήρ για ένα λεπτό από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, Προστασίας Καταναλωτών και Δημοσίου. Ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια ήταν πολύ καλή η συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πολύ καλό δρόμο για να πετύχει το στόχο της του 20% συμμετοχή στον ΑΠΕ ε, στο ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2020. Στην ψήξη και τη θέρμανση γίνονται μεγάλες πρόοδοι, αλλά λείπει μια πρόταση για τις μεταφορές. Γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια επενδύσεων για την παραγωγή βιολογικών καυσίμων περιμένω μια νέα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μετά το 2020 ε, και ε, να δώσει πιο ε, σταθερή προοπτική σε εκείνους που παράγουν βιοκαύσιμα. Λυπάμαι που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ ο θετικός ρόλος των δασών. πόσο σημαντικό είναι η συμμετοχή του δάσους ε, στο μείγμα αυτό των βιολογικών καυσίμων. Γιατί υποτιμούμε τη γεωργία και τη δασοκομεία. Θα μπορούσε ε, να δημιουργήσει 146.000 μόνιμες θέσεις εργασίας ο κλάδος και 162.000 εποχικές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για την Επιτροπή ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο κύριος Σαμαζή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η COP21 κατέδειξε το θεμελιώδη ρόλο των περιφερειών και των πόλεων για τη μετάβαση προς ε, κοινωνίες με χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Για τη δική μας Επιτροπή Ρέγγι τα κονδύλια από τα ταμεία συνοχής μπορούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δική μας Επιτροπή λοιπόν Περιφερειακής Ανάπτυξης εκφράζει τη λύπη της που η κινητοποίηση αυτών των κονδυλίων ήταν από 1,1% το την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και έφτασε στο 1,4% στην τρέχουσα 2014-2020. Γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση σε δήμους και περιφέρειες στην Ευρώπη να κινητοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και να ανασκουμποθούν. Ιδιαίτερα οι πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες θα πρέπει να θέσουν ε, το φιλόδοξο στόχο τη ενεργειακή αυτονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μαρζή. Δεν βλέπω τον κύριο Μπόκοβιτ στην αίθουσα, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Λίζε για ένα λεπτό εξ ονόματο Επιτροπή ε, Περιβάλλοντο. Για την έκθεση Πίπερ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίπερ και όλους όσους ε, το βοήθησαν για να ε, καταθέσει την έκθεση και βλέπουμε πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ και ΕΝΔΗ. Θέλουμε ευελιξία. Θέλουμε ευελιξία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα μέτρα του άρθρου 5. Χρειαζόμαστε ασφάλεια σχεδιασμού σε σημαντικά κομμάτια τη οδηγία, όχι μόνο μέχρι το 2030, αλλά και πέρα από αυτό. Και μεγάλε συζητήσει γίνονται και στι δύο επιτροπέ. Έγιναν μάλλον και στι δύο επιτροπέ για τον απότερο στόχο εμείς υποστηρίξαμε με πλειοψηφία όχι υπέρ του 40%. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω την, ε, το συμβιβασμό που κατέθεσε το ΕΛΚ. Υποστηρίξαμε το 40% αλλά δεν θεωρώ ότι αποτελεί ρεαλιστικό στόχο. Αλλά τουλάχιστον 30% ζητάει το ΕΛΚ. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνονται συζητήσεις για το κατά πόσο θα πρέπει να ξεπεραστεί το 20% στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενδεχομένω και ο κύριος Γιούγκερ να μην το υποστηρίζει αυτό. Αλλά ο κύριος Γιούγκερ υποσχέθηκε στις αρχές της θετίας πριν την εκλογή του να ξεπεράσει αυτό το 20% και θα πρέπει να τηρήσει αυτές τις υποσχέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Λίζα και τώρα εξ ονόματος των ομάδων θα ακούσουμε τους ομιλητές. Δύο λεπτά ο κύριος Μπέντσεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας πω για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει στο μέτωπο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, ε, ενεργεία, συγγνώμη, ευχαριστούμε την κυρία Μπερμέχο για τη συνεργασία. Ε, οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές. Υπήρχαν κάποιες διαφορές μεταξύ μας αλλά οι στόχοι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να επιτευχθούν. Νομίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επίσης συμφώνησαν για αυτούς τους στόχους και δεσμεύτηκαν σχετικά. Υπάρχει ο στρατιωτικός στόχος του 2030. Αξέπαινε αυτή η προσπάθεια. Ελπίζω ότι θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και θα πρέπει ο τη της εφορίας να θυμόμαστε όλα αυτά. Και για να νιώσουμε τις πηγές ενέργειας επίσης είναι σημαντική η στόχη για το ενεργειακό μείγμα που θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία επασχόληση. Οπότε θα πρέπει να βρεθούν κάποιε λύσει μακρόπνοε, να δημιουργηθούν κατάλληλε συνθήκε στην αγορά. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τις ε, εταιρείε και τους καταναλωτές. Θα πρέπει, σύμφωνα τις αρμοδιατές τους, τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν. Θα πρέπει να θεσπίσουν και κάποιες ενισχύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που δεν τις κρίνουμε ρεαλιστικές αλλά κάποιες άλλες είναι λογικές. Νομίζω... Σας ευχαριστώ συνάδελφε Μπέντσαν και τώρα το συνάδελφο έχει... Το λόγο έχει ο συνάδελφος Πόκο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίπερ για την εξαιρετική συνεργασία για την ε, έκθεση, για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η τρέχουσα οδηγία αποτελεί μια καλή βάση για την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων στα πλαίσια και του COP21, αλλά μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς μόνο εφόσον ε, επιλύσουμε κάποια προβλήματα της οδηγίας. Υπάρχει υπερβολική ευελιξία και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν ε, πετυχαίνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, γιατί αν δεν αλλάξει τίποτε, δεν θα πετύχουμε τους στόχους της μείωσης του 20% μέχρι το 2020. Νομίζω ότι οι βουλευτές στα πλαίσια της Επιτροπής Βιομηχανίας επεσήμεναν ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, μεγαλύτερη εφαρμογή. Σε ό,τι αφορά το 40% τώρα, είμαι πεπισμένος ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει στεναρά να υποστηρίξει αυτόν τον στόχο. Γιατί αν είπα να χωρίσουμε ε, έναντι του 40% ουσιαστικά λέμε ότι δεν θέλουμε, ότι αποδεχόμαστε ότι θα είμαστε ανεξάρτητοι σε ό,τι αφορά τα ρηκτά καύσιμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα της ενεργειακής αποβατικότητας δεν το είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη οδηγία. Το συζητάμε τώρα και χαίρομαι. Και εδώ πέρα λοιπόν γίνεται μια έκκληση προς τα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει να κάνουν μια θετική έναρξη και αφετηρία στο θέμα αυτό σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 και σε ό,τι αφορά τα σχέδια των κριτών μελών για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τέλο, το ζήτημα των ε, λοιπόν κανονισμών που επηρεάζουν το θέμα αυτό. Συζητάμε το θέμα του ETS, τη εμπορία ρήπων, το οποίο σχετίζεται ασφαλώ ε, πολύ με το θέμα αυτό και υπάρχουν μεγάλε αλληλεπικαλύψει. Αντί να υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των νομοθετημάτων αυτών, θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι συμπληρωματικά το ένα προ το άλλο. Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό το γεγονό. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μα ε, καταθέσει αποτελεσματικέ λύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πούχα. Επιτρέπετε μπλε κάρτα του κυρίου Χριστοφόρου, κύριε Πόχε. Παρακαλώ κύριε Χριστοφόρου. Κύριε, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτέ τι μέρε πραγματικά είμαι προβληματισμένο κατά πόσον η κλιματολογικη και περιβαλλοντολογική στοχή είναι ταυτόσιμοι και με του ενεργειακού. Επικεντρωνόμαστε μόνο στα θέματα ενέργεια ενώ το περιβάλλον κινδυνεύει. Και επειδή η πατρίδα μου αυτή. Παρακαλώ, άλλαξε μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένο ότι η κλιματική περιβαλλοντολογική στόχη είναι ταυτόσιμοι με του ενεργειακού. Δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στα ενεργειακά θέματα και να αφήνουμε έξω το περιβάλλον. Και επειδή η πατρίδα μου αυτέ τι μέρε υπέστη μια άνευ προηγουμένου οικολογική περιβαλλοντολογική καταστροφή από ανεξέλεκτε πυρκαγιέ, με αποτέλεσμα να χαθούν και ανθρώπινε ζωέ δασοπυροσβεστών που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει... Excuse me, excuse me. Συγγνώμη. Ε, γαλάζια κάρτα είναι αυτή. Ερώτηση πρέπει να κάνετε στον ομιλητή. But you have only... Ναι, έχετε μόνο 30 δεύτερα για το σκοπό αυτό, τα οποία και έχετε υπερβεί. Please. Επικεντρωνόμενο σε αυτό πρέπει να πω Μικρόφωνο. Μικρόφωνο, παρακαλώ πώς μπορούμε εμείς να κινητοποιήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ταμεία αλλά και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους, ώστε μαζί με τους ενεργειακούς στόχους να υλοποιούμε και τους περιβαλλοντολογικούς και να μπορούμε να προστατεύουμε τα δάση μας αλλά και να τα αποκαθιστούμε όταν υφίστανται ζημιές όπω έγινε αυτή τη στιγμή με την Κύπρο και ανέφερα το θέμα αυτό και νομίζω ότι το ανέφερε και ο Επίτροπος, αν δεν κάνω λάθος. Ένα κομμάτι της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και αυτός ο δεσμευτικός στόχος του 40% είναι αυτός που θα συμβάλλει για την μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ. Αν και δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον αυτό συνδέεται με την Κύπρο απαραίτητα, για να είμαι ειλικρινής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόχα. Ένα λεπτό. Η κυρία Φανβοσέιτ Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, σήμερα ψηφίζουμε δύο σημαντικές ενεργειακές εκθέσεις. Η μία έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση και η άλλη με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα κράτη-μέλη συμφωνούν για τους στόχους ε, που θέλουν να πετύχουν. Ε, απειλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως να βάλει πολύ ψηλούς και μη ρεαλιστικούς στόχους. Από τη μια θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, μειώσουμε την χρήση ενέργειας. Υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν η μισή ενέργειά μας χάνεται, μάλλον πηγαίνει στη θέρμανση και στη ψήξη, αλλά χάνεται γιατί κυριολεκτικά φεύγει από πόρτες και παράθυρα σε πρώτο λόγο θα πρέπει να ποντάρουμε στην ενεργειακή απόδοση, αλλά να μπορεί και ο πολίτης να βλέπει τις επενδύσεις να είναι προς δικό του όφελος. Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουμε στόχους ρεαλιστικούς και όχι ανεδαφικούς. Να είμαστε φιλόδοξοι, δεν λέω, αλλά να παραμένουμε και ρεαλιστικοί. η ε, δεσμευτική εθνική στόχη λοιπόν δεν είναι ρεαλιστική που ζητάει ο συγητής. Είναι γεγονός ε, ότι ε, θα πρέπει κάποια κράτη-μέλη να κοιτάξουν και πέρα από τα σύνορά τους για να επιτύχουν τους στόχους. Τότε γιατί ζητάμε υποχρεωτικούς και δεσμευτικούς εθνικούς στόχους σας. Έχουμε ευρωπαϊκή προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαν για 1,5 λεπτό το λέει έχει και ο συνάδελφος κ. Γερπράντη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και θα ήθελα να ξεκινήσω ε, αναφέροντας δύο ενεργειακές εκθέσεις οι οποίες πρόσφατα δημοσιεύτηκαν. Η πρώτη, ένα άρθρο αναφέρει ότι η ολική και η ε, ηλιακή ενέργεια ε, καταστρέφουν τα ορεικτά καύσιμα και μιλάει για το 2015 ότι το ΑΠΕ ήταν διπλάσια από τα ορεικτά καύσιμα και χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρθηκαν project στο Μεξικό και αλλού όπου ε, εφαρμόστηκαν ε, προγράμματα ΑΠΕ επειδή ήταν πιο φτηνά. Και η άλλη έκθεση αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει την φήμη της ως ηγέτης σε ενεργειακά ζητήματα και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Πέρσι οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, μειώθηκαν κατά 21% ενώ οι δαπάνε στον υπόλοιπο κόσμο στον τομέα αυτό ε, γνώρισαν έκρηξη. Αυτό αναφέρει η έκθεση και μας ανησυχεί αυτό. Και αυτό που βλέπουμε στον κόσμο είναι μια παγκόσμια αύξηση και μια παγκόσμια ζήτηση για ε, φθηνέ και αξιόπιστες πηγές ενέργειας, όπως είναι οι ανανεώσιμες. Και είναι επίσης ε, καθαρές οι ανανεώσιμες. Αυτό είναι μια υπέροχη παραπλευρή συνέπεια Άρα, χρειαζόμαστε βασικά φτηνή και αξιόπιστη ενέργεια. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιαστούμε και να επικεντρωθούμε στι ΑΠΕ. Το πιο βλαβερό θα ήταν ο συντερτισμό εδώ. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επικέντρωση με φιλόδοξου δεσμευτικού στόχου. Και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταρτίζει τις εκθέσεις, τις προτάσεις της το Σεπτέμβριο, να καταθέσει φιλόδοξους δεσμευτικούς στόχους. Δεν είμαι βέβαιος, λέει ο Πρόεδρος, αν ο συνάδελφος πίσω στην αίθουσα αν ε, επιτρέπετε μπλε κάρτα και ερώτηση από έναν συνάδελφο του οποίου το όνομα δεν μπορώ να εντοπίσω αυτή τη στιγμή. Μίκο. Ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες ότι δηλαδή χρειάζεται νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο και επίση το Nord Stream 2 είναι ένα έργο το οποίο προχωρά και η καγκελάριος Μέρκελ το έχει εγκρίνει. Δεν σημαίνει αυτό το ότι ε, τελικά ίσως τα όνειρά μας ε, δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ θα πρέπει να το πάρουμε σε σοβαρά την υπόθεση γιατί αλλιώς να σταματήσουμε μιλάμε για ένα νιώσιμο Yes. Chairman, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Δεν νομίζω ότι το Nord Stream είναι μια καλή ιδέα. Αλλά αυτό που ακόμα περισσότερο ε, με ανησυχεί είναι ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει επιβραδυνθεί η υπόθεση Τη Ενεργειακή Ένωση. Έχουμε 28 χωριστές αγορέ. Θα πρέπει αυτή την ε, μετάβαση προ ασφαλή, καθαρή ενέργεια ε, να, την αγκαλιάσουν αυτή την ιδέα. Αυτό θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Πρόεδρος. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπενίτο Σιλουάγα. Καλημέρα σα, κυρίε και κύριοι. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Πριν μιλήσουμε για ενέργεια θέλω να πω ότι είναι μεγάλη έκπληξη που σας βλέπουμε εδώ στην Ολομέλεια στην ίδια Ολομέλεια όπου είστε τόσο ακριβοθόρητος όπου η Μεγάλη Συμμαχία σας επιτρέπουν να εξηγείτε γιατί το όνομά σας συνέχεια φαίνεται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής. Μας έχει συνηθίσει όμως το κόμμα σας αυτά τα πράγματα. Την άλλη φορά που θα έρθετε εδώ στην Ελομέλεια, κάντε μας τη χάρη να έρθετε να μας ε, δώσετε λόγο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις ε, που σας ζητούν οι πολιτικές ομάδες. Γιατί να έρχεστε και κλεισμένων των θυρών με ε, γνωστές ερωτήσεις δεν διαλύει καμία αμφιβολία. Ευτυχώς που την Κυριακή θα κάνουμε ένα βήμα στις εκλογές στην Ισπανία για να έρθουν στα πράγματα άνθρωποι χωρίς κουνιάδους με ε, ενεργειακά θέματα και χωρίς λογαριασμούς ε, στον Παναμά. Έλεγα λοιπόν ότι η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να είναι ε, δεσμευτική υποχρέωση για όλα τα κράτη-μέλη και προτεραιότητα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια οδηγία για τις ανανεώσιμες με πλαίσιο σταθερό και που να τις ευνοεί. Σε αντίθεση με αυτά που κάνει η χώρα μου η κυβέρνησή της με τα θέματα της ηλιακής ενέργειας. Χρειαζόμαστε δημοκρατική ανανέωση όσο και μετα... ενεργειακή μετάβαση στην Ισπανία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπενίτο Σιλουάγα. Θέλω να διακόψω λίγο τη συζήτηση και να καλωσορίσω ε, την πρώτη ομάδα επισκεπτών.